89, 90, 91 ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές εγκρίνεται. 97. «92, 93, 94 ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, αποχές ελέγχουμε 92, 93, 94 ανοίγει η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας ψηφοφορίας το ΕΛΚ ζήτησε πολλά η Γκουε α η ΓΚΟΕ μπορεί να αφαιρέσει ένα και το ΕΛΚ δύο Περιμένουμε την ΚΟΕ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Α, για τραβήξτε το. Πέρες ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 18 κατά εγκρίνεται. 95 ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 2, 97, ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά, αποχές, απορρίπτεται. 96, ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά, αποχές, απορρίπτεται. 98, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβασμός 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ενβι 20. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ε, κάνετε μαζί. Ψήφι υπέρ. Κατά τον 8 και τον 9 και τον 11 ψηφικά κατά να το ελέγξουμε αρχίζει η ψηφοφορία 107, 8, 9 τον 11 ψηφίσατε όλοι εντάξει πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται Συμβιβασμός 3. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. 1-1-5 προσήκη στο 3 ψήφι υπέρ. Αποχές απορρίπτεται. 20 εισηγητής ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1-3-5 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 1-3-6 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25 έμβη ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1-3-7 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1-26 Ένβη, ένβη, με συγχωρείτε, ψήφι υπέρ. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Περίεργο είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος. 30, 39, 140 και δύο μαζί ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 138 καταπτύπη, 141 ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, αποχές απορρίπτεται. 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 143 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 146 σαράντα έξι ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 145 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 147 και 148 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 149 εισηγητής ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 152 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 τη Επιτροπής Περιβάλλοντος, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 154, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 150, 151, 153, από κοινού, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 155-156 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Επιτροπή περιβάλλοντος 30 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 157 υπέρ κατά αποχές Έμβη MV31 καταπίπτει και περνάμε στην 158 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 159 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται με 162, 163, 165 μαζί. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. NV32. Να για να ελέγξουμε. 161, 2, 3, 5. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Α, απορριπτεται MB32, those in favor. 168 υπέρ κατά απορρίπτεται. 168 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23 αποσύρεται. 161, 164, 166 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 160, 167 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 169 ψήφοι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 170 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 24. 172 μαζί ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Επιτροπή Περιβάλλοντος 28 καταπίπτει. 171 καταπίπτει. με τώρα στο 175, 76, 77 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές μπορούμε να ελέγξουμε. 75, 76, 77. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορία Απορρίπτεται. 25, 179, Επιτροπή Περιβάλλοντος 33. Από κοινού ψηφίζουμε ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 174, 180 ψήφι περ κατά αποχές εγκρίνεται. 173, 78, 82 ψήφι υπέρ. Κατά. Συγγνώμη, συγγνώμη, έχει ήδη καταπέσει. Ωραία. Η 181 της κυρίας Φώστε, ψήφι υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. MV34, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 183 και 184 ψήφι υπέρ κατά αποχές μπορούμε να ελέγξουμε την 183 και 184 αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Συμβιβασμός 4. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 5. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 6. Άρθρο 7. Η ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. NB46 NB46 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2-5-3 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Από 9 2-5-6 της κυρίας Φώστερ ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. Και τα υπόλοιπα καταπίπτουν. Περνάμε στο συμβιβασμό 7. Συμβιβασμός 7. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 8. Άρθρο 11. Συμφωνούς 8. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36. Με το 2, 7, 8. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το 2, 7, 4, καταπίπτει. 38. 2, 7, 8 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στο άρθρο 16. 2,79 και 2,80 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράτημα 1, 2, 8 2 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 281, 283 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ένβι 49 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ένβι 50 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2, 8, 4, 5, 6 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. εγκρίνεται. 52 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε την MP52, ε, αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας και απορρίπτεται. 2-8-7 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. MB53 ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές απορρίπτεται. MV54 ψήφι υπέρ. Κατά. 55 ψήφι υπέρ. Κατά. το 55, το 55 να δούμε. Πέρας ψηφοφορίας. MV56 ψήφι πέρα Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Κοιτάξτε, μας ενοχλεί ε, το τηλεφώνημα που κάνετε. Είτε τελειώστε με το τηλεφώνημα, είτε βγείτε εκτός ε, τροπολογια 291, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Όλες καταπίπτουν. Περνάμε τώρα στο 2.95 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 40, τροπολογία 40. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμβη 57 κατά πίπτη παράρτημα 2 ψηφιπέ 3 09 ψηφιπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμβη 61 ψηφιπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 ψηφιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 307 κατά πίπτη και το 311. Περνάμε στο MV62 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 313 <coughs> ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 64 από την άλλη ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 65 Έμβη υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. All those in favor. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η τελική παράγραφος τώρα με τη σειρά η πρώτη του εισηγητού, έχουμε και εδώ και την πρώτη τροπολογία του εισηγητού, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ένβη, παριθμόν 1, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 50, 51 και 53 είναι υπέρ κατά θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο, ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 52 του κυρίου Μαρινέσκου, πήνε είναι υπέρ, πήνε κατά, αποχές, απορρίπτονται. Ένβη, παριθμόν 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 54, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ένβη ε, 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ένβη 4 υπέρ κατά αποχέ, απορρίπτεται. ενβι 5 υπέρ κατά αποχέ, απορρίπτεται. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Υπέρ κατά απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ένβη 9 υπέρ κατά Ένβη 9 και πάλι υπέρ ευχαριστώ κατά αποχές εγκρίνεται. Ένβη 10 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την nv παριμών 10 ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρα πάμε στην 5 και 63 υπέρ. 5 και 63 υπέρ. Ερκατά. Εγκρίνεται. 64 και 68 υπέρ κατά αποχές Απο... εγκρίνεται και τώρα πάμε στην ένβη παριθμών 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται, 72 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ε, Ένβη, 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 9 και η 74 πήγαινε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 73 καταπίπτει, 77 είναι υπέρ, είναι κατά, αποχές, απορρίπτονται. 78 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Ένβη 15 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος της ε, NV15 ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ένβη. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτω. Τελική ψηφοφορία για την νομοθετική πρόταση όπως έχει τροποποιηθεί. Ψηφίζουμε. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά δύο εποχές και τώρα για το δημοκρατικό ψήφισμα ψηφίζουμε ψήφισαν όλοι πέρας εγκρίνεται 33 υπέρ 10 κατά και μία εποχή συγχαρητήρια κύριε Λάχτφριντ πάει το ένα τώρα Κάτι μου λέει ότι θα είναι τα πράγματα από τώρα και στο εξή κάπως πιο δύσκολα, λέει ο πρόεδρος. Και πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω στο σχέδιο της έκθεσης για το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στους κοινού κανόνες για την κατανομή των χρονοθυρίδων στα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Γιος Ουτζιάς είναι ο εισηγητής μας. Ξεκινούμε από την 16 του εισηγητού. Ποι είναι υπέρ, ποι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, 90 και 91. Υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτωτα 92. Υπέρ κατά αποχές έλεγχος για το 92 ψηφίζουμε ψήφισαν όλοι πέρασε εγκρίνεται 94 είναι το επόμενο που είναι υπέρ είναι κατά, αποχές, κρίνεται. 1795 και 96 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική 1. Υπέρ κατά αποχές. Έλεγχος για την συμβαστική υπαρχμόν 1. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφορίας απορρίπτεται και τώρα πάμε στην 104 που είναι υπέρ που είναι κατά αποχές απορρίπτεται καλά να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο κατά τη δική μου γνώμη 4 προς 1 ήταν η αναλογία των ψήφων υπέρ και κατά ψήφισαν όλοι ε, μιλούμε για την 104 τώρα. Εκεί βρισκόμαστε. Ψήφισαν όλοι. Είναι η πρώτη μετά από την συμβαστική. Γιατί κατέπεσε η συμβαστική. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεν κρίνεται. Τι να σας πω, κρίνω από αυτά που βλέπω, από όσους σηκώνετε τα χέρια. 99, καταπίπτει. 199 για το άρθρο 9 παράγραφος 8 που είναι υπέρ και είναι κατά άλλη μια φορά υπέρ κατά αποχές έλεγχος μιλούμε για το 199 δεύτερη σελίδα. Το λέει ο σοσιαλιστές αυτό. Έτσι. Θα ήθελα να πω στους συναδελφούς ότι επειδή κατέβησε ο συμβασμός θα πρέπει να ψηφίσουμε για όλες ε, τις ε, τροπολογίες οι οποίες είναι στο κομμάτι του κειμένου που έχει τον γκρίζο γκριζοπό χρωματισμό. Άρα μιλούμε τώρα για το 199 έρχεται από τους καλούς φίλους μας Φιντάντζα και Καντσιάν. Έχουν όλοι ψηφίσει. Όχι, δεν νομίζω από ό,τι βλέπω εδώ. Πέρασε ο φορείας. Εγκρίνεται. πάμε τώρα στο 100 89 της κυρίας Σερακιάνη. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για το 189 επίσης της κυρίας Σερακιάνη. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ο φορείος. πάντως το 206 μέχρι και την 213. 206 213 213 είναι υπέρ. Είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα στο 79. Εκεί θα πάμε, θα ψηφίσουμε τους ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την τροπολογία υπαριθμών 11 ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 75. Υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 218, 219, 220. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 228. Ε, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκλίνεται. Συγγνώμη, εγκρίνεται, εγκρίνεται, διορθώνει ο πρόεδρος. Να σας πω ποιο είναι το θέμα. Το ότι δεν ψηφίζεται κατά ε, ομάδα πολιτική, αλλά επί τη βάση της εθνικής προέλευσης. Αυτό είναι το θέμα. Όχι, εγώ είπα ποτέ, ποτέ δεν ψηφίσω ε, σαν ε, Άγγλος. αυτά ήταν οι 222 και τώρα 295 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αυτό μέχρι 299. 300, 301, 302. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, τον Όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό, πρόεδρος. Πού είμαστε. Α, στο 68, Ρικέ. Υπέρ κατά αποχές. Έλεγχος για το 68. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. ροκή πλουσιδία 69, Κύριε Λίχτεμπεργκερ. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Γίνει έλεγχος. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αυτό ανατρέπει την, στο ε, ε, συμβασμό. Αν πάτε 106 ποιο είναι υπέρ. Και είναι κατά. Αποχές. Μάλλον βρείτε αλλά θα κάνουμε τελικό έλεγχο για 105 και 106. Ψηφίζουμε. Σηκώστε τα χέρια σας να φαίνονται πέρα ψηφορίας και όντως απορρίπτονται. 107 υπέρ. 107 υπέρ. Κατά. να Απορρίπτεται. 108. Ντεμπάκερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 109. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική υπερθμόν 2. Για να δούμε την πίσω αυτή το πάει καλύτερα. Περ, κατά. Α, αποχές εγκρίνεται. Άρα πάμε στο 180. Συγγνώμη, 128. 128. Πίνε υπέρ. Είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 129. Υπέρ. Κατά αποχές, έλεγχος. Για το, το 29 ψηφίζουμε. Πέρας. Οριακά εγκρίνεται. 130 κυρίες Φώστερ, υπέρ. Κατά. Α, αποχές, έλεγχος. Γιατί είμαστε τόσο κουρασμένοι, ποτέ δεν ξέρει κανεί, οπότε ξαναψηφίζουμε ηλεκτρονικά για το 130. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Είκοσι δύο. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Σαφής πλειοψηφία εδώ. Σάσολια. 28 Περκατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά αποχές κάνουμε έλεγχο για το 135 ψηφίζουμε ψήφισαν όλοι πέρας Απολύτως. 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 136 υπέρ κατά Εγκρίνεται. 24. Υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Εκατόν σαράντα. Υπέρ. Κατά. όχι. Έλεγχος για το 140. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 25 του εισηγητού. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 138 ως προσθήκη 25 υπέρ κατά εγκρίνεται κατά καταπίπτει, οπότε πάμε τώρα στο 26 του εισηγητού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. το 26. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά, αποχές. 32. υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 159 υπέρ. Κατά. Νομίζω απορρίπτεται, αλλά θα κάνουμε έλεγχο. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Με μερική πλειοψηφία εγκρίνεται. Πέρ. κατά Αποχέ. έλεγχος για το 160. Ψηφίζουμε. ακόμη πιο η πλειοψηφία εδώ πέρα, με ένα ψήφο. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για το 162. Καλά θα περάσουμε στην Ολομέλεια. Το βλέπω. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται και αυτή. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για το 33. Ψηφίζουμε. Πέρασε ευφορίας. Ένας παράπονα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Γκάλερ. Πέρας. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Απόχευση. Ελέγχο για το 34 ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι υπέρ. Και εγκρίνεται αυτή. 163. Υπέρ. Κατά. Αποχές αν σε και το 63. Παρακαλώ. Ο... Ε, ψηφίζουμε τώρα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτονται. 35. Ε, του εισηγητού υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Μου φαίνεται ότι το κάνουμε όλα ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. 164. Φιντάντσα. Ψηφίζουμε κατευθείαν ηλεκτρονικά τώρα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 178 now. 178 τώρα. Υπέρ. Κατά. Οχές. Έλεγχα το 178. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι πέρας. Εγκρίνεται. 179. Υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Εγκρίνεται. 171 λοιπόν, για το 191 θα κάνουμε τώρα έλεγχο. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 182 καταπίπτει. έλεγχο για το 182. 183, έλεγχος. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. και 185, συγγνώμη, ο πρώτος 182. 182 σας όλοι υπέρ, κατά, εποχές, έλεγχος του 182, ψηφίζουμε, ψήφισαν όλοι, πέρας, απορρίπτεται, και τώρα, 185 από κοινού, υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος, και για αυτά τα δύο ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Τα οποία καλά μέχρι τώρα και τώρα πάμε 186, κύριο που υπέρ κατά, εγκρίνεται 187 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος για το 187, ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 188. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχο 188. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. συγγνώμη, εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 201 απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτονται 280 σας όλοι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 203 κατά αποχές εγκρίνεται 204 και 205 204 και 5 λοιπόν εγκρίνονται 214 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 215 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 217 υπέρ, κατά, αποχές. Εργασία για το 217 ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρες. Απορρίπτεται. 229 και 230 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 231 και 232 υπέρ. Κατά. Αποχές. κρίνονται, 233 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 294 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 230 30 36 υπέρ κατά αποχές Ευρωπαϊκός έλεγχος για το 236 πέρασε. ισοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. από το ΕΛΚ περισσεύει ένας. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Η 235 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 237 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Άποχες Εγκρίνεται. Και έτσι περνάμε στην 248. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 40 του σύγητου. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 249 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. σεμπιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και έτσι περνάμε στην 272. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 273, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 274, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 274. Να το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορία. Αν ψήφισατε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 275. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και πάλι στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ έναρξη ψηφοφορία για την 275. Αν ψηφίσατε όλοι, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Η 276 υπέρ, κατά, αποχές. Να το ελέγξουμε για την 276 παρακαλώ έναρξη ψηφοφορίας. Αν ψηφίσατε όλοι, πέρας, όχι ακόμη. Τώρα. Απορρίπτεται. 277 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε, αν και νομίζω ότι είναι ίδιο το αποτέλεσμα, ψηφίζουμε για την 277 παρακαλώ. Αν ψηφίσετε όλοι. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Πέρασε τις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 278. είναι κύριε Γκρό. Ε, ο κύριο Τεβέρεκα, ο 278 υπέρ κατά αποχέ Να ελέγξουμε το 278 παρακαλώ, ενάξη πληροφορία. Αν ψηφίσετε όλοι και αν ψήφισε σωστά και ο κύριο Γκρό. πέρας ψηφοφορία. απορρίπτεται. 279 υπέρ. Κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας ελέγξουμε και για την 279 παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Αν ψήφισατε όλοι, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται όντως. Οριακά. 280 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε την 280 παρακαλώ, έναρξη ψηφοφορίας. Αν ψηφίσατε όλοι, Πέρας. Εγκρίνεται. 281 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 282 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 282. Έναρξη ψηφοφορίας. Μα δεν έχουμε αρχίσει καν την ψηφοφορία για τις υπηρεσίες αντάφους. Μην παραπονιέστε. 282, λοιπόν, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 303, υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε την 303, Έναξη ψηφοφορίας. Αν ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 304 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Αλλά ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Είναι ψηφοφορία για 304. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Εγώ είμαι σχετικά βέβαιος, αλλά άμα δεν συμφωνούν και οι μισοί βουλευτέ. 305. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές να το ελέγξουμε παρακαλώ. Να ελέγξουμε τη 46. Ένα ψηφοφορία. Αν ψηφίσετε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Για τη 45 ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορία. Αν ψήφισετε όλοι. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. απόχέ Εγκρίνεται. Η 49 υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την 49 ένεξη ψηφοφορίας. Αν ψηφίσετε όλοι, πέρας. Απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 50 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την 54. Ένας ψηφορίας. Πολύ αμφιβάλλω, αλλά αν ψήφισατε όλοι, ολοκληρώνεται η ψηφοφορία. 27 υπέρ, 17 κατά, εγκρίνεται. 54, 55 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 4 υπέρ. Α, συγγνώμη, έχει καταπέσει. Στην 5 πάμε λοιπόν. 5 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται 60 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται η 6 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται 61 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται 62 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται 64 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, 7. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 63. Υπέρ. Α, όχι. Δεν έχει καταπέσει 63. Θα είχε καταπέσει αν είχε εγκριθεί 64. Αλλά πρέπει να την ψηφίσουμε τώρα. 63. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε, να το ελέγξουμε αν θέλετε ηλεκτρονικά. Έναξη ε, ψηφοφορία για την 63. Αν ψηφίσετε όλοι, ολοκληρώνει την ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Η 9 κατά 5. 65 καταπίπτει. Στη 10 πάμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Η 81. 81 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος ηλεκτρονικός παρακαλώ για την 81. Ένα της ψηφορίας. Αν ψήφισατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Η 82. Έχει αποσυρθεί 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την 83 αν ψηφίσατε όλοι. της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην άλλη σελίδα. Την 86. 86. Υπέρ. Κατά. Τα Αποχές εγκρίνεται. 87. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 88 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ την 88. Έναρξη ψηφοφορία. νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά ας το ελέγξουμε, γιατί τα χέρια σας κουράζονται όλο και πιο πολύ. Αν ψηφίσατε λοιπόν όλοι, πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται οριακά. Α, συγγνώμη. Ισοψηφία. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ή 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για την ε, νομοθετική πρόταση όπως έχει τροποποιηθεί. Έναρξη ψηφοφορίας παρακαλώ. Αν ψηφίσατε όλοι, ολοκληρώνει την ψηφοφορία. εγκρίνεται 39 ψήφοι υπέρ, 5 κατά, καμία αποχή και τώρα σε ό,τι αφορά το νομοθετικό ψήφισμα ψηφίζουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά αν ψηφίσατε όλοι ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία εγκρίνεται με το ίδιο αποτέλεσμα 39 ψήφοι υπέρ 5 κατά συγχαρητήρια στον κύριο Ούτζιας και καλή τύχη σας ευχόμαστε για την Ολομέλεια Άντε, ψηφίσαμε λοιπόν δύο εκθέσεις. Μιας, θα σας πρέπει να ενημερώσω ότι ε, θα φύγω και ο κύριος Γκάλερ είναι το άτομο που έχω επιλέξει. Είναι ο εκτός για να ψηφίσει στη θέση μου. Κοιτάξτε, όσο εφόσον πάρετε μαζί την κάρτα ψηφοφορία σας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.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 ο κατάλογος ε, παρατήματος 1α ε, για τον κατάλογο των ε, διαγραφών ποιότητας. Θα ακολουθήσει τη διατύπωση της τροπολογίας 52, όπως αναφέρεται στη διατύπωση της τροπολογίας 52. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα, πρόταση κανονισμού για τις υπηρεσίες εδάφους, στα αεροδρόμια της Ένωσης και κατάργηση της οδηγιας 96 46-67. Ξεκινάμε με τις τροπολογίες 53, 54, 55, 57 που είναι για απόρριψη της πρότασης υπέρ κατά άποχες. Αυτά πρέπει να το ελέγξουμε όπως και να έχει. Έναρξη ψηφοφορίας παρακαλώ. Αν ψηφίσετε όλοι, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 22 ψήφι υπέρ, 20 κατά. So that brings us to the end of the, the voting on the handling. Και έτσι δεν ψηφίζουμε λοιπόν. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για τις υπηρεσίες εδάφους με 22 ψήφους υπέρ, 20 κατά. 22 ψήφοι υπέρ, 20 κατά. Ως εκ τούτου εγκρίνεται και έτσι ε, απορρίπτεται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 να σας πω ότι μπορεί να μην προβλήθηκε στις ε, οθόνες, αλλά ήταν 22 ψήφοι υπέρ και 20 κατά. Πιστέψτε με. Και de facto, επειδή πλέον δεν έχουμε κοιτάξει το τρίτο νομοθετικό κείμενο, να σας υπενθυμίσω ότι δεν υπάρχει πλέον πακέτο και ότι έχουμε πλέον ε, χαλάσει το πακέτο και τώρα η απόρριψη θα περάσει στην Ολομέλεια, θα πρέπει να ε, επικυρωθεί από την Ολομέλεια. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία της έκθεσης της κυρίας Wills για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης. Ας ψηφίσουμε παρακαλώ. Εντάξει. Right, we start with the, again, it's uh, amendment. Η τροπολογία υπαριθμών 1. Πρόκειται για την οδηγία του Συμβουλίου για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρηση. Τροπολογία υπαριθμών 1 και πάλι προτείνει απόρριψη τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Άρα περνάμε στην ε, ψηφοφορία. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Ξανά, ξανά. Η 19. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 31 και 15 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 33 ως προστίκη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 17, 34 και 52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 Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Η 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ την 47 ηλεκτρονικά. Έναρξη της ψηφοφορίας. Αν ψηφίσετε όλοι, Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 51. 50 συγγνώμη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οι δύο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τρία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τέσσερα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η δέκα. Το κ. σαν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται η 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε την 11 παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές Ας ελέγξουμε και τη 13 παρακαλώ έναξη ηλεκτρονική ψηφοφορίας αν ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 16 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 39 ψήφοι υπέρ, μία κατά, τέσσερις αποχές. Συγχαρητήρια στην κυρία Wills. Εγκρίνεται. To your members if there is doubts about the no, we'll send it to them anyway. Can I just, um, members? Συνάδελφοι, επειδή ήταν οριακή η απόρριψη της πρότασης για um, τις υπηρεσίας εδάφους. Θα την εκτυπώσω και θα σας την στείλω για να ξέρετε ποιο ήταν το ακριβές αποτέλεσμα. 44, 44 ε, βουλευτές ψήφισαν, 22 υπέρ, 20 κατά, 2 αποχές. Αν θέλετε λοιπόν θα σας στείλουμε τις λεπτομέρειες. Στο επόμενο σημείο της ημερής της διάταξης, στις 5 προβλέπετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή που δείξατε κατά τη διάρκεια της ευφορίας. We'll have a 10 minute break λεπτά διάλειμμα μέχρι τις 4.30 παρακαλώ. Στις 4.30 ξεκινάμε την έκθεση Fleckenstein και μετά την πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. κύριε Φλάκισταν, κατάφερα να συγκεντρώσω μερικά μέλη, γιατί τα καταφέραμε και χθες δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Φλάκισταν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. δεν έχει αλλάξει τίποτα επί το περιεχομένου και βρισκόμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο που βρισκόμασταν. Και άρα μπορώ να σας πω ότι χαιρετίζω το συμβαστικό, τη συμβαστική πρόταση. Ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχαν στην εξέβριση του συμβιβασμού και ότι είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην εφαρμογή. Εγώ θεωρώ ότι δεν χρειάζεται και δεν χρειάζονται και οι πολυάριθμοι συνάδελφοι που βρίσκονται εδώ να ακούσουν εκ νέου τα ίδια επιχειρήματα. Σας ευχαριστώ και, πάλι για την καλή συνεργασία. Και σας ευχαριστώ τώρα κύριε Τουμπλάντζη για το ΕΛΚΑ. Ναι, Πρόεδρε. Μια μου πιέζει ο χρόνος να σας τα πω ε, σύντομα να εξευχαριστήσω τον, τον εισηγητή και πάλι για, για τη στάση του, για τη συνεργασία μας. Ήταν πάρα πολύ εύκολο να επικοινωνήσουμε για αυτό το θέμα για το οποίο μπορέσαμε να βρούμε πολλούς κοινού τόπους και σύμφωνα σε πολλά σημεία, οπότε το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ θετικό, πάρα πολύ καλό για όλους και για όλο το κοινοβούλιο και φυσικά για την ε, καταθάλασσα ασφάλεια. ανασφάλεια. Η κυρία Μπιλμπάου. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Βέβαια και εγώ δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις προσπάθειες που κατέβαλε αυτές εξ αρχής, ούτως ώστε να μπορούμε να συζητήσουμε όλες αυτές τις τροπολογίες. Αρκετά συνεργαστήκαμε και είναι η ικανοποιημένη πολιτική μας ομάδα για τις συνθήκες οι οποίες περιέβαλαν αυτή τη συμφωνία. Βέβαια θα θέλαμε να συμφωνήσουμε ακόμα περισσότερο σε ακόμα περισσότερα πράγματα, αλλά πάντως ε, νομίζω ότι τελικά από την πίεση του χρόνου θα αναβαθμίσουμε τις δυνάμεις μας και θα μπορέσουμε να, να, να κάνουμε αυτά που δεν μπορέσαμε μέχρι σήμερα να κάνουμε. Και φυσικά τροχοπέδι είναι από τα κρατημέλη της προγραφιές μας και βέβαια εν κατακλείδη να ευχαριστήσω για όλες αυτές τις προσπάθειες της Κομισιόν και του Συμβουλίου με όλες αυτές τις τροπολογίες που αφορούν στο άρθρο 5. Έχουμε την διατύπωση, αλλά έχουμε και το άρθρο 11 και σας ευχαριστώ. Thank you very much, Eva. I don't know whether you want to say anything for the Greens or, or Jackie. Do you want to say anything? Ήρθε στην για τους Πρασίνους, Jackie για το ECR, λέει ο Πρόεδρος. Ε, ε, ούτε η Κομισιόν θα πει τίποτα και σας υπενθυμίζω ε, τα σχετικά με το, με το ότι στις 25 Δεκάτου είχαμε στην Ολομέλεια την ανακοίνωση των θέσεων Συμβουλίου και, και Κομισιών και έγινε επομένω κατά αυτόν τον τρόπο η πρώτη συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση και η προθεσμία είναι η 8η ενδεκάτου το μεσημέρι για τις τροπολογίες και στις 27 ενδεκάτου θα γίνει η ψηφορία στην ε, Επιτροπή και ελπίζουμε το θέμα να πάει το Δεκέμβριο στην Ολομέλεια. Καλώς, ωραία, επομένω αν δεν έχετε καμία ένσταση ε, κλείσαμε αυτό το θέμα και τώρα πρέπει να περιμένουμε τον κύριο Κεμάλ, Καμάλ όσον αφορά ε, την έκθεση του ανταγωνισμού στις 5 ανεμένα τον έρθει οπότε άρα, άρα Πάμε για τις 5 ώρες, που να τελειώσουμε τις 5.30. Άρα, αναμονή, δεκάλεπτος και συνεχίζουμε μετά. Α, αυτά γίνονται όταν απορρίπτονται κάποιες ε, προτάσεις και δεν κρατάει όσο πρέπει. Το δύο ώρα που προβλέπει την ψηφοφορία. Hey, colleagues, we'll start again. First... συνόδελφοι, ξαναρχίζουμε πρώτα-πρώτα. Κύριε Καμάλη, με το οποίο που ήρθατε. Είμαι βέβαιος ότι σας είπανε ότι θα έπρεπε να ψηφίσουμε περισσότερη ώρα, αλλά τέλος πάντων τελειώσαμε πιο νωρίς. Ευχαριστούμε που ήρθατε στις 5 η ώρα. Είναι μεγάλη υπόθεση για μας. Τώρα μιλούμε για την έκθεση που αφορά το σχέδιο της νομοδότησης για ε, την πολιτική του ανταγωνισμού. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καμάλ με μεγάλη μου χαρά ντεμπουτάρω σήμερα στην Επιτροπή. Ευχαριστώ και για την θερμή υποδοχή. Ε, και δεν θεωρώ ότι είναι προσωπικό, προσωπικό και ύβρι προ το πρόσωπο μου το ότι ήρθαν λίγοι συνέλθει, Δεν πειράζει. Δεν ξέρω τι έγινε πριν έρθω, οπότε καλύτερα να είμαι προσεκτικό και επομένω καλύτερα να προσέξω τα πρώτα μου βηματάκια σε αυτή την Επιτροπή, τα παρθενικά. Οπότε είναι βασικό ότι θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι τα κράτη-μέλη συνεχίζουν την πορεία προ αυτή την ε, μια από την ανταγωνισμού είναι λάβουν υπόψη το διαχωρισμό ε, δημοσίου και, και ιδιωτικού τομέα και πολλές φορές το πρόβλημα είναι η θέση των κρατών μελών, πολλές φορές είναι θέμα εφαρμογής, πολλές φορές θα πρέπει πριν ε, προχωρήσουμε σε ένα νομοθέτημα να λάβουν υπόψη το τι ήδη ισχύει. Έχουμε μια συνθήκη με τις ΗΠΑ και προσπαθούμε έτσι να δούμε τι, τι κάνουν εκεί, τι κάνουν οι Αμερικανοί συμμαχοί μας και βέβαια από μια μεριά έχουμε ε, ανταγωνισμό. Τέλος πάντων, ε, ε, εγώ ήμουν έτοιμος να συμμετάσχω ε, αφελώς και ορεξάντας στη θέση μέτρων για τα αεροδρόμια. Τέλος πάντων, πέραν των όσων έγιναν πριν έρθω εδώ, έχω να σας πω ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα της, ε, των, δυνατοτήτων, των παραγικών δυνατοτήτων. Ε, ξέρετε ότι η τουζερή συζήτηση ε, σε συγκεκριμένη περιοχή σχεδόν της των αεροδρομίων στη χώρα μου και βέβαια αυτό το θέμα δεν αφορά με τη μου χώρα αλλά και με τις νέες αγορές. Πολλές χώρες της και το ίδιο ζήτημα. Να σας πω τώρα. Εμεί θέλουμε όσο να έρθουν περισσότεροι φραγμοί και να γίνει καλύτερη εφαρμογή. Και όσον αφορά τι ε, μεταφορέ των αυτοκινητόδρομων και επίση. Κοιτάξτε, όταν κάνει ρίξει μια ματιά στη δέσμη των για του λιμένε, βλέπει κανεί τι πρέπει να γίνει όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση σε διάφορα κράτη-μέλη. Και πολλέ φορέ, αυτό που μου λένε ότι ο κόσμος θέλει περισσότερη προσδοτώ προς τον προς τη φιλοσοφία της αγοράς. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινηθεί προς το να ανοίξουν οι ιστορικές υπηρεσίες στο εσωτερικό και γενικότερα στις μεταφορές να υπάρχει πιο υγιής ανταγωνισμός και από την άλλη μεριά έχουμε προβληματισμό των τοπικών κοινοτήτων για κάποια περιβαλλοντικά θέματα. Πάντως, βασικά, αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε την υπάρχουσα νομοθεσία, αλλά να εφαρμόζεται καλύτερα. Γιατί κάποιο του καίει ακριβώ το θέμα τη ορθή εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού. Εδώ λοιπόν θα βάλω τελεία, τόσο ώστε να μπορέσουν να μιλήσουν και άλλοι για το θέμα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ΕΛΚ τώρα. Σας κύριε ε, συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Όχι, δεν είναι δύσκολο κανείς να συμφωνήσει με τα όσα είπατε, με τα όσα προτείνατε. Ε, βεβαίως ε, αντιλαμβάνομαι ότι λόγω του χρόνου και της διαθεσής σας δεν μπορέσατε να πείτε περισσότερα. Τέλος πάντων, αυτά τα οποία διατυπώνετε στο έγγραφο είναι πάρα πολύ θετικά. Οπότε εμείς εύκολα σας δίνουμε το πράσινο φως. Σήμερα πάντως για τον ανταγωνισμό είναι μέρα θλιβερή, ε, αναμφισβήτητα και θα πρέπει ακριβώς όπως γίνεται και για, για τους ε, βασιλιάδες λέμε ο βασιλιάς πέθανε, ζήτω το βασιλιάς ε, και αυτό ισχύει για την εσωτερική αγορά, σύμφωνα με τόσα έγιναν και με κάθε σεβασμό ε, σε σχέση με αυτούς που έχουν την αντίθετη άποψη. Νομίζω επομένω ότι σήμερα δεν, δεν μας τιμά αυτό το οποίο έγινε, ούτε αυτό το οποίο έχει γίνει, τιμά την ελεύθερη αγορά. Θα συνεχίσουμε επομένω την πορεία μας προς την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς για τις μεταφορές και κατά αυτόν τον τρόπο επίσης θα πρέπει να έχουμε εγγυήσεις με μια δικαίωση όρων ανταγωνισμού και για δυτικό και για δημόσιο τομέα, οπότε καθ' αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να ισχύσουν όλα αυτά και στον τομέα των μεταφορών. Γιατί για όλη την οικονομία είναι πάρα πολύ σημαντικοί οι μεταφορές από τις οικοδομές ε, του κατασκευαστικού τομέα μέχρι τη γεωργία. Επομένω, πρόκειται για κάτι σαν ε, φαινόμενο της, της ε, που διακρίνει τη σχέση ε, των μεταφορών με τους άλλους οικονομικούς τομείς. Τώρα πρέπει να σας ε, πω το ότι προβλέπει νέα δέσμη για τα αεροδρόμια και για τα αεροσλημένες μέχρι το 2013 και θέλουμε επομένω η Κομισιόν να δείξει θάρρος. Γιατί αυτό το θέμα εκρεμεί εδώ για πολύ καιρό. Και σας υπενθυμίζω ότι οι εξαγωγές μας γίνονται από τους λιμένες το να εφαρμοστούν οι κοινοί κανόνε, οι κανόνε για την ανάπαυση, οι κανόνε για την εργασία σε κάθε ε, τρόπο μεταφορά είναι κάτι το απαραίτητο ώστε να έχουμε ελεύθερο ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα σε σχέση με τα περιφερειακά αεροδρόμια είναι θετικό το ότι η Ευρωπαϊκή ε, ε, Επιτροπή θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το τι γίνεται και λέμε τώρα για την απότερη περιφέρεια, γιατί για τους νήσους, γιατί εκεί για να λειτουργήσουν οι λιμένες πρέπει να δούμε τι, πόσο μπορεί να καλύψει να βοηθήσει ο δημόσιο τομέα. Αυτό αφορά και το περιφερειακό αεροδρόμιο, μεσαία κατηγορία, ενδιάμεση τέλο πάντων. Ε, να δούμε τι θα γίνει σχέση με τις, με τις ενισχύσεις. Εμείς πάντως είμαστε υπέρ κάθε μέτρου που οδηγούν σε απελευθέρωση όλων των τρόπων μεταφοράς γιατί όλα αυτά έχουν σημασία για την οικονομία, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Και ταυτόχρονα επίση θα πρέπει παρεχθούν, να έχουμε κάποιε εγγυήσει, ώστε να κατοχυρθούν τα δικαιώματα των ε, επιβατών και να υπάρχουν ε, άρτιε, σωστέ, ποιοτικέ υπηρεσίες, Τικάου, για τους σοσιαλιστάς. Θα πρέπει και εγώ να ευχαριστήσω, να συγχαρώ τον εισηγητή και να ξεκινήσω μια ερώτηση. Ποια ήταν τα θετικά στοιχεία, οι θετικέ επιπτώσει ε, της σταδιακής, ε, του σταδιακού ανοίγματο σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό καταρχάς για τους επιβάτες, για τους εργαζόμενους και θα ήθελα να θέσω να αναφέρω και τις επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει επίσης να ε, τις εξετάσουμε. Θεωρώ ότι αν θέλουμε πραγματικά μια ενιαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόμαστε και σωστό ανταγωνισμό. Και στην περίπτωση αυτή χρειαζόμαστε μια ε, υποδομή σε, άλλ, σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί σήμερα υπάρχουν πολλές διαφορές στην ανάπτυξη των υποδομών στα μεμονωμένα κράτη-μέλη και γι' αυτό θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να επενδύσουμε στον εξυγχρονισμό των σχετικών υποδομών, των ε, συστημάτων μεταφορών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά και τις χώρες που προσχώρησαν το 2004. Επίσης, θεωρώ ότι είναι σημαντικό για να υπάρχει ε, σωστός και δίκαιος ανταγωνισμός στον ιστορικό, στην ιστορική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να άρουμε τα εμπόδια για την ε, ε, ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων. Θεωρώ ότι η άρση των εμποδίων σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους και την κινητικότητά τους είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να ε, δραστηριοποιηθούμε πιο έντονα σε ό,τι αφορά τέλος την εφαρμογή του συστήματος αυτού στον συνδρομικό κλάδο, έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε, δυστυχώς. Και στην τελική ανάλυση διαπιστώνω ότι δεν έχουμε επαρκή αρμοδιότητα. Μόνο στις οδικές μεταφορές, κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ ε, της πλήρους απελευθέρωσης του συστήματος Καμποτάς και μέχρι το 2014 θα υποβληθεί σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ε, σχετική οδηγία σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση του Καμποτάς. Δεν ε, είναι πραγματικά ενοποιημένη η ενιαία αγορά και αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα κρατήσεων και αγοράς εισιτηρίων πολύ λειτουργικό. Υπάρχουν λοιπόν πολλά εμπόδια ακόμα για τους επιβάτες σε ό,τι αφορά τα ταξίδια που θέλουν να κάνουν. Χρειαζόμαστε λοιπόν πιο πολύ διαλειτουργικότητα. Και εδώ διαπιστώνουμε ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναλύει ουσιαστικά θέματα ανταγωνισμού από πλευράς μεταφορών, αλλά δυστυχώ δεν καταδεικνύει τις επιπτώσεις του ανταγωνισμού στα μεμονωμένα τμήματα, στους μεμονωμένους τρόπους μεταφορών σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις υποδομές κτλ. Θεωρώ λοιπόν ότι με την χρονομοδότηση ε, αυτή θα πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αυτούς τους διαφορου... διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των τρόπων μεταφοράς, ε, τη διαλειτουργικότητα, την σταδιακή, το σταδιακό άνοιγμα των αγορών και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και στους επιβάτες αλλά και στις επιχειρήσεις, στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αυτά λοιπόν από πλευράς μου. Θα ήθελα όμως να θέσω και ένα άλλο ερώτημα, το εξής. Τι επιπτώσεις έχει αυτή η πολιτική ανταγωνισμού σε ό,τι αφορά τις διεθνείς σχέσεις, γιατί ξέρουμε ότι στον τομέα των αερομεταφορών αλλά και στις οδικές μεταφορές υπάρχουν, εξακολουθούν μάλιστα να υπάρχουν ορισμένα εμπόδια σε ό,τι αφορά τις μεταφορές. Υπάρχουν ε, και διεθνείς συμβάσεις στον τομέα αυτά θα πρέπει να έχουμε λοιπόν υπόψη να ακριβώ αυτέ τι διεθνεί σχέσει, τι ε, ε, συμβάσει που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτε χώρε και ποιε είναι οι επιπτώσει αυτών στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Επόμενο ομιλητή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και να πω ότι συμφωνώ με τον τρόπο προσέγγισης του. Το πρώτο είναι ότι με ικανοποίησε ότι είναι υπέρ αυτού του πακέτου των ε, αεροδρομίων. Η επίγεια εξυπηρέτηση δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα φιλόδοξο, έτσι ώστε να μετακινηθούμε σε μια πιο ε, ανταγωνιστική βιομηχανία την παροχή περισσότερων ανταγωνιστικών ε, ε, υπηρεσιών. Η Επιτροπή δεν ήταν ε, ιδιαίτερα φιλόδοξη και από την άλλη πλευρά το Κοινοβούλιο δεν όθησε προς σωστή κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά τη χωρητικότητα των αεροδρομίων, αυτός είναι ένας τομέας που με βρίσκει απέναντι στον εισηγητή. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο χωρητικότητας στην Ευρώπη και το πρόβλημα θα έλεγα ότι εντοπίζεται, είναι εντοπισμένη αυτή η έλλειψη χωρητικότητας. Και ένα από τα θέματα που θα πρέπει να εξετάσουμε είναι το πώς να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη χωρητικότητα πριν να αρχίσουμε να επεκτηνόμαστε. Νομίζω ότι είναι σκόπιμο να δούμε τι κάνει η Λουφτκάνησα στη Γερμανία με το επωνομαζόμενο multi-hobbing, να εξετάσουμε το αεροδρόμιο του Μπέρμιχαμ που είναι περίπου το ίδιο. Έχει κάποιο mini hub και το συνδέει με το, και συνδέεται με το Λονδίνο. Νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό και στην Ευρώπη, όπου υπάρχει μία έλλειψη χωρητικότητας Εκεί που υπάρχει, υπάρχουν τρένα υψηλής ταχύτητας και θα μπορούσαν να κάνουν πολύ καλά την ε, δουλειά. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα τρένα και να αντικαταστήσουμε πάρα πολλές ε, μικρές ε, πτήσεις και τα αεροδρόμια να έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα για άλλες πτήσεις. Νομίζω ότι αυτό το θέμα της χωρητικότητας σηκώνει περισσότερο σκέψη. Γιατί το ζητούμενο είναι να τη χρησιμοποιήσουμε καλύτερη. Το να ζητάμε διαρκώς μεγαλύτερη χωρητικότητα και από άποψη υπερβαντική είναι λανθασμένο. Θα ήθελα να αναφερθώ στο τελευταίο σημείο που αφορά τον τομέα των σιδηροδρόμων. Χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο στον τομέα αυτό. πακέτο των σιδηροδρόμων δεν είναι το ίδιο και με το, με το πακέτο των αεροδρομίων. Αυτό είναι κάτι που όλοι θα μπορούσαμε να στηρίξουμε. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη πρόσβαση έτσι ώστε να υπάρξει μια πιο ανταγωνιστική είναι πιο ανταγωνιστική σιδηρόδρομη. Διαφορετικά οι τιμές θα αυξάνονται συνέχεια για τον καταναλωτή. Και αυτό δεν βοηθάει επουδενή την ανταγωνιστικότητά μας. Ένα καλό σιδηρόδρομος θα μπορούσε να δώσει τις κατάλληλες υποδομές για να κινηθεί όλη η οικονομία. Σε ένα σωστό πλαίσιο λοιπόν θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε κάτι καλύτερο. Και πραγματικά Περιμένω τη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών για να δούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να το προωθήσουμε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριο Κράμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή. Υποστηρίζω κυρίω την προσέγγιση του. Λέει ότι χρειάζεται μια προσέγγιση η οποία θα προσανατολίζεται στην αγορά. Έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά απέχουμε παρασάγκα από το στόχο αυτό. Δεν έχουμε κανένα ανταγωνισμό. Είναι μη ναι, δίκαιος ανταγωνισμός και επιβαρύνεται τελικά το κλίμα. Και αν ναι, χρειαζόμουν ένα μάρτυρα, θα ανέφερα τον Ιωάννη Λούντεβικ, ο οποίος στη Γερμανία είπε ότι στον τομέα των μεταφορών δεν υπάρχει κανένα ανταγωνισμό στην Ευρώπη. Να σας πω και προσθέτω ότι είναι η χειρότερη κοινωνική, κοινωνικός προγραμματισμός που τελικά ε, είναι ε, βλαβερός για το περιβάλλον. Κάποια παραδείγματα να σας δώσω. Δεν έχουμε τους ίδιους ε, κανόνες. Θα πρέπει είτε να πληρώνουν όλοι τους ίδιο τον ίδιο είτε όχι. Αλλά οι αερομεταφορές, οι αεροπορικές εταιρείες δεν το πληρώζουν. και οι συνδρομικές εταιρείες το πληρώνουν. Ή θα πρέπει να τα πληρώνουν όλοι, είτε όχι. Είτε θα πρέπει να ενταχθούν όλοι στον εμπόριο ρήπων, είτε όχι. Αλλά οι αεροπορικέ εταιρείε εξαιρούνται. Στις οδικές μεταφορέ το ίδιο συμβαίνει. Ζητήσαμε ε, διότι για τα τρένα. Ενώ στους δρόμους ισχύει το ότι κάθε κρατος μέλος επιβάλλει ότι επιθυμεί μόνο φορτηγά, μόνο φορτηγά μέχρι 12 τόνους, ε, με περιορισμούς για να μην ε, ε, θίξουμε και τους Ελβετούς. Και στις πλωτές οδούς το ίδιο συμβαίνει. Οι τιμές είναι ελεύθερες. Και μπορώ να συνεχίσω. Αυτό λοιπόν είναι τρελό, κοιτώντας τι γίνεται με τις αεροπορικές εταιρείε. στη Γερμανία, να σα πω τουλάχιστον, στον Ντόρτμουντ, στο Κάσελ, διατηρούνται αερολιμένες όπου γίνονται δύο πτήσει την ημέρα μόνο. Και η επιχειρηματολογία είναι ότι, κοιτάξτε, επενδύσαμε για τα αεροδρόμια αυτά, να συνεχίσουμε να λειτουργούν. Αυτά είναι τρελό, είναι παλαβό. Θα πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση για την Ryanair, το ανέφερα ήδη. Η Ryanair αναφέρει ότι έχει 500 ε, εκατομμύρια ευρώ ως κέρδος τα τελευταία χρόνια. Αλλά έχουν ε, και ζημία 300 εκατομμύρια. Από πού προκύπτει όμως ε, αυτό το παράδοξο ότι έχουν επιδοτήσεις που τις πληρώνουν οι Ευρωπαίοι προλογούμενοι. Τεράστια λοιπόν αυτή η φούσκα, όπως η φούσκα των ακίνητων στην Ισπανία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσανατολιστούμε στην αγορά. Θα πρέπει να προσανατολιστούμε σε τέτοιες άρχες. Να συμπεριληφθεί και το εξωτερικό κόστος. Εδώ και χρόνια κατηγορώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ξέρετε αυτό. Ξέρετε πως έχει η κατάσταση εδώ και χρόνια και δεν κάνετε τίποτα. Ε, αντιμετωπίζετε τμηματικά τις μεταφορές, όχι όμως το σύνολο του τομέα, για τον ε, ανταγωνισμό. Ανταγωνισμός, ναι, αλλά όχι εξίσωση στους ίδιους μισθούς dumping και θα πρέπει να καταλάβουν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κρατημέλη ότι δεν θέλουμε τον ανταγωνισμό του dumping. Ε, δεν θα δούμε που ισχύουν οι πιο χαμηλοί μισθοί. Όχι, θα πρέπει να υπάρχουν και κοινωνικές ρήτρες. Όχι έτσι. Μία πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι Γάλλοι έχουν ναι, εισάγει το rolling Stock tax ε, στις σιδηροδρόμους σε ό,τι αφορά την κατάργηση του επιχειρηματικού φόρου. Και τώρα τι γίνεται. Για τους Γάλλους δεν αλλάζει τίποτα, αλλά για αυτούς ε, που είναι εξωτερικοί, εξωτερικές εταιρείε πληρώνουν διπλό φόρο και στη χώρα τους και στη Γαλλία. Και εδώ και δύο χρόνια προσπαθούμε κάτι να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητούμε κάτι να γίνει. Αλλά δεν κάνετε τίποτα. Αποδέχεστε ότι είναι μη δίκαιο ο ανταγωνισμός. Τι κάνετε όμως. Θα σας δώσουμε το λόγο σε λίγο και πραγματικά υπομονώ να μάθω αν θα κάνετε, αν ποτέ να κάνετε κάτι για αυτά. Ο κύριος Κούμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εφόσον έχουμε έναν εμπειρογνώμονα μαζί μας ε, για θέματα πολιτικής ανταγωνισμούς και σε ό,τι αφορά και την ε, ετήσια έκθεση, μπορούμε να θέσουμε μία σειρά ερωτημάτων προς τον κύριο Καμάλ. Στην Επιτροπή σας ε, συζητιέται η οδηγία για την παραχώρηση. Και εκεί συζητιούνται θέματα όπως το τι είναι κριτικές υποδομές ε, για την διατήρηση ε, ε, των λειτουργιών μιας κοινότητας ενός κράτους. Και βλέπουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να συνεχίσει να απονέμεται με διαγωνισμού στο μέλλον. Εκεί κάπως δημιουργούνται αμφιβολίες, για παράδειγμα η υδροδότηση κτλ τα θέματα μεταφορών, υγειονομική περίθαλψη, να το σημειώσουμε αυτό. Αν αυτά, αυτές οι υποδομές ε, αφαιθούν στα χέρια καπιταλιστικών ε, μονάδων και προσθεθούν για παράδειγμα και τα νοσοκομεία και τα υπόλοιπα, πάντα θα πρέπει να υπάρχει απόδοση 6-7%. παραμένουμε ανοιχτοί. Δεν χρειάζεται όλοι να αγοράσουμε ελληνικές, ελληνικά ομόλογα. Αλλά θα ήθελα ως εμπρεγνώμονας να μας πείτε πού θεωρείτε ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να μην καταλήξουμε σε ένα ξέφρενο καπιταλισμό, σε μια ξέφρενη απελευθέρωση προκειμένου να υπάρχει και το δημόσιο χέρι, το οποίο θα ορίζει, κοίταξε να δεις, αυτό είναι υποχρέωσή σου. Είτε βγάζει κέρδο είτε όχι. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η λεπτή ισορροπία να τηρηθεί. Ίσως, ε, Πρόεδρε, σήμερα που έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω, ήθελα να το θίξω αυτό το θέμα, το θέμα της αρχής. Ο Πρόεδρος. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Κέλλα, πρωτού δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα με τις μεταφορές και την εσωτερική αγορά και αν πιστεύετε στο Θεό υπάρχει εσωτερική αγορά. και αυτό σε σχέση με άλλους τομείς όπως ε, οι τηλεπικοινωνίες. Ενδεχομένως υπάρχουν ε, λόγοι, αλλά ενδεχομένως σε ορισμένες περιπτώσεις είναι θέμα μονοπωλίων. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Αλλά υπάρχουν τομείς και νομίζω ότι ο Μάκρη έχει δίκιο. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τις μεταφορές στα πλαίσια της Επιτροπής της Πολιτικής Ανταγωνισμού. Εγώ δεν θα έλεγα να αναφερθούμε σε συγκεκριμένους τομείς που υπάρχουν προβλήματα. Συνεχίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών, να βρισκόμαστε αντιμέτωποι. με ναυτιλιακές εταιρείε που θέλουν να μεταφέρουν προϊόντα από το Λίβερπουλ, στο Πάρι, από το Αμβούργο, στη Γένοβα και θα πρέπει να συμπληρώσουν διασαφήσεις ε, τελωνιακές ή ε, άλλες. Η εσωτερική αγορά είναι καλαμπούρι, είναι αστείο. Δηλαδή, αν θέλετε να μεταφέρετε αγαθά από τη μία χώρα μέλος στην άλλη, θα πρέπει να συμπληρώσετε μία σειρά από έντυπα. Δεν ξέρω, ας πούμε, συμβαίνει θα συνέβαινε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι εσωτερικό όμως. Θα πρέπει λοιπόν να λυθεί αυτό το θέμα. Θα πρέπει να αναπτύξουμε τις λεωφόρους, τις θάλασσες, όλες αυτές τις μεθόδους. Όταν κοιτάξετε τον τομέα των αερομεταφορών, ένας άλλο τομέας, ανοίγουμε τον ανταγωνισμό, ανοίγουμε την αγορά το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε τις διάφορες εταιρείες τύπου Ryanair, οι οποίες έχουν μπει στην αγορά. Δεν λέω ότι είμαι κατά αυτού. Θα πρέπει να πω ότι είμαι κατά μερικών από τις πρακτικές που συνεχίζονται. Και μία από αυτές αφορά το θέμα της μίσθωσης αεροσκαφών. Τζάκι μπορεί να επιβεβαιώσει ότι λόγω αυτού του συστήματος δεν υπάρχει ανταγωνισμός πλέον στην πτήση Manchester Places. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός στο Manchester Παρίσι ε, σαρδεγκολα Τώρα τα πάντα τα καλύπτουν οι, οι, οι Brussels Αυτό το σύστημα της συνεργασίας σκοτώνει τον ανταγωνισμό. Δεν φαίνεται να δραστηριοποιούμεθα κατά αυτού του τύπου ε, συνεργασίας. Στη μια εσωτερική αγορά βεβαίως, βεβαίως θα πρέπει να έχουμε αυτές τις μεθοδεύσεις Μόλις ε, ανοίξετε το καμποτάσι στην ακτοπλοεία και στον τομέα αυτό, όλοι θα τρελαθούν και θα, λέ, θα αρχίσουν ε, να λένε ότι μπαίνουν στο περιθώριο, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία. Γιατί θα πούνε, γιατί αφήνετε τους μεταφορείς ε, από την Πολωνία να καλύψουν αυτό το, το κενό. Συνεπώς, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί θα αρχίσουν και πάλι οι αγρότες να εξεγείρονται. Να κοιτάξουμε τώρα το θέμα των σιδηροδρομικών μεταφορών. Θα πρέπει να γίνει κάποια πρόοδος στο τομέα της αγοράς. Αυτό είναι το τελευταίο οχυρό θα λέγαμε που έχουμε και υπάρχει κάποια κίνηση, αλλά χρειάζονται βοήθεια, χρειάζονται κάποια αρρωγή για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πρέπει να ανοίξει η αγορά δίχως να δοθεί μια μορφή σε βοήθεια για να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι κλασικό αυτό με την ε, αγορά των σιδηροδρόμων. Θα πρέπει όμως να κάνουμε βήματα μπροστά. Ένα τελευταίο σημείο ότι έχουμε ένα σύστημα, είτε μας αρέσει είτε όχι, υπάρχει ένα σύστημα φορολόγηση. Εγώ δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες. Έχουμε ένα σύστημα που επιτρέπει στη μία χώρα ε, μέλος να επιβάλλει φόρους σε άτομα που φεύγουν από τη χώρα αυτή, ενώ σε άλλες χώρες δεν υφίσταται αυτό και υπάρχει ένα σύστημα που επιτρέπει σε ορισμένες χώρες να αυξάνουν τις τιμές ε, των καυσίμων ενώ άλλες όχι. Ενώ έχετε υπάρχουν, επιβάλλονται φόροι σε μία χώρα και όχι σε άλλη, σε μία άλλη, τότε ε, οι συνολικές παροχές ε, θίγονται άμεσα. Κάτι θα πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά τη φορολογία, έτσι ώστε όλοι να κινούνται στο ίδιο επίπεδο. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν ορισμένες χώρες μέρη που είναι λίγο πιο ευαίσθητες σε σχέση με άλλες. Αυτή όμως είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ε, δεν μπορείτε να κινηθείτε έτσι όταν όλα τα ε, παρόλες ανομαλίες που υπάρχουν στον τομέα της ακτοπλοείας, ε, των αεροπορικών μεταφορών, των σιδηροδρομικών μεταφορών. Επιτροπή. Η Επιτροπή. Τέρι Μπρόμς. Ε, α, Τέρι, εσείς, μάλιστα. Α, Τέρι, μου αρέσει πολύ αυτό το όνομα. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που μας περιμένετε να έρθουμε και να συμμετάσχουμε στη συζήτηση γιατί αυτό αποδεικνύει το πόσο σημαντικό είναι το σημερινό ζήτημα και θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή γιατί είναι πάρα πολύ αξιόλογο το σχέδιο του κειμένου, θέτει πολλά σημαντικά ζητήματα και συμφωνούμε 100% μαζί του και με ένα σωρό βουλευτές που ήδη έχουν πει ότι προβληματίζονται γιατί είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό το πώς θα πετύχουμε να υλοποιήσουμε και στις μεταφορές σε ενιαία αγορά και επίσης ε, ε, το θέμα είναι το ότι θα πρέπει για τα καράτη μελη να λάβουν τις ευθύνες τους και λαμβάνω υπόψη όλη αυτή τη σειρά των προτάσεων, των συστάσεων που ακούσαμε σήμερα. Όσον αφορά αυτό το οποίο ρωτήσατε, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο να σχολιάσουμε όσον αφορά κάθε αυτό το σχέδιο του κειμένου. Συνεχίζονται φυσικά όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές, ε, οι συζητήσεις, τις υπηρεσίες μας και για το καμποτάζ και ελπίζουμε ότι είναι το χρόνο και στα πλαίσια που έχουν τεθεί θα είμαστε έτοιμοι. Πάντως νομίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποκτήσει περισσότερη πλήρηση τώρα το πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Ασχολούνται με αυτό περισσότερες από μία ε, ε, ε θα πρέπει επομένως από τι πλευρές ταυτόχρονα δούμε το ζήτημα και Ξέρετε, έχουμε επιταχύνει τους ρυθμούς με τους οποίους ασχολούμε με τα θέματα ε, της ε, Συνεργαζόμαστε και με την αρμόδια γενική διεύθυνση για τις αγορές και όλοι μαζί προσπαθούμε επομένω να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ε, ε, γύψουμε στα τμήματα της ενιαίας αγοράς. Δεν τόσο καλά όπως είναι οι μεταφορές. Και γι' αυτό επομένω προσπαθούμε να επιτύχουμε τη συνεργασία μεταξύ των επιμέρου των διευθύνσεων και να μπορέσουμε και στι μεταφορέ να υλοποιήσουμε την ενιαία αγορά. Να δούμε και εμεί που είμαστε η Γενική Διεύθυνση του Ανταγωνισμού πώ μπορούμε και εμεί να βάλουμε το λιθαράκι μα για όλη αυτή την υπόθεση. Θα μακρύσω ο δρόμο που έχουμε διανύσει και ελπίζουμε ότι τώρα πια ο κόσμος έχει δει το θέμα πολλές διαφορετικές απόψεις, λοιπόν μπορούμε να συνθέσουμε και να προχωρήσουμε με αυτή την ετησία έκθεση για να διαπιστώσουμε τι απομένει για να γίνει και σε επίπεδο μελών και να δούμε και εμείς με τη σειρά μα, αν είναι ανταγωνισμό πώς μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε για τι μεταφορέ. Α, θα κάνετε την ετησία έκθεση. Πολύ καλό. Τι θα κάνετε όμως για τον αθέμητο ανταγωνισμό. Είδατε τι κάνουν οι Γάλλοι. Δύο χρόνια τώρα δεν κάνουν ε, ε, διαδρομές ε, χερσαίες πέρα από τα σύνορά τους. Τι γίνεται. Θα κάνετε τίποτα, Επιτροπή. Ναι, λαμβάνετε υπόψη αυτό το οποίο είπατε. Δεν είμαι εγώ η εμπειρογνώμων ε, για το θέμα των μεταφορά. Θα πρέπει να το συζητήσουμε με του ειδικού συναδέλφου και να δω πώ είναι η κατάσταση. Και σα δίνω το λόγο μου ότι θα σα ε, αναφέρω σχετικώ. Πρόεδρο ναι. Ε, υπάρχει αυτό το θέμα των κοινών πτήσεων και ξέρουμε ότι αυτό καπνίγει τον ανταγωνισμό. Ιδίως σε συγκεκριμένες διαδρομές. Αυτό είναι ακριβώ και το πρόβλημα. Είναι καθημερινό το πρόβλημα. Και αλλού και στη δική μου χώρα έχει εξαλειφθεί, εξαφανιστεί ο ανταγωνισμός. Άρα θα πρέπει κανείς να εφαρμόσει σωστά τα όσα ισχύουν πριν πει πάμε να κάνουμε ενιαία αγορά. Και ο Μάγκλ, αυτό ήθελα να σας πει, φαντάζομαι. Καμάλ. Στην παρθενική μου εδώ εμφάνιση, πρέπει να σας πω ότι θεώρησα πολύ ενδιαφέρουσα τη συζήτηση. Θα λάβω υπόψη όλα όσα εθίγησαν. Πάντως νομίζω ότι όλοι θέλουν να υπάρχει ενία αγορά όσο πιο σύντομα γίνεται. Και πάντα κάθε αλλαγή θα πρέπει να δικαιολογείται, να αιτιολογείται. Ο κύριος Μπαρνιέ, ο αρμόδιος επίτροπος, έχει, θέλει να προχωρήσει προς την ε, ενιαία αγορά της μεταφορές. Και εμείς να κάνουμε μέσα ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνει αυτό. Και ό,τι δεν λειτουργεί εύρυθμα, να το διορθώσουμε όσον αφορά τις ε, μεταφορές. Πάντως δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι θα πρέπει να δούμε και αντίκτυπο που έχουν όλα αυτά για τους εργαζόμενους. Ναι, για τα περιφερειακά αεροδρόμια και τα δίκαια. Και ε, στη χώρα μας ισχύει το ίδιο. Πάντως με το Επιτροπή Μεταφορών εσείς θα πρέπει όσοι και όσοι να αποφασίσετε σε μια τέτοια έκθεση για τον ανταγωνισμό πόσο θέλετε να μπούμε στις λεπτομέρειες. Και άπαξ και να αποφασίσουμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε προς μια τέτοια δεύτερη πράξη στο έργο της ολοκλήρωσης της ζωικής αγοράς να δούμε ποιους συγκεκριμένου τομεί θέλουμε να προωθήσουμε για ολοκλήρωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και περιμένω πώς και πώς την εργασία μου στους κοιόδους συγκεκριτές. Ευχαριστώ κύριε Καμάλ. Να λέει από τα δεσμένες μέχρι τώρα δεν είχαμε κάνει, δεν είχαμε απορρίψει τίποτα μέχρι σήμερα. Δηλαδή, οπότε να, συνήθως δεν κάνουμε κάτι τέτοιο. προθεσμία για τις τροπολογίες 13 ε, Δεκάτου, ψήφος στις 18 ε, Δεκάτου στην Επιτροπή και στην Οικονομική θα γίνει η ψήφιση τον Ιανουάριο και θα πάει 13 επομένως του μηνός και 18 Δεκεμβρίου η ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω με τίποτα άλλο θα δει τίποτα άλλο τίποτα διάφορα. Οπότε δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω του ε, διερμηνεί για τη δουλειά του και του ε, συναδέλφου και κυρίω τη λήξη τη